Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα θέμα στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης σε αυτήν την δημόσια κρόαση. Λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερες συνθήκες μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συναντήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Τζόναθαν Χιλ. Εγώ προσωπικά εκτίμησα όλους ιδιαίτερα την ευαισθησία που επέδειξε αποφασίζοντας να παραιτηθεί μετά από το δημοψήφισμα αυτό. όλοι οι συντονιστές ομόφωνα ε, ξέφρασαν τα αισθήματά τους. Είπαν ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά μαζί του αυτά τα χρόνια που ήταν υπεύθυνο επίτροπος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, υπηρεσίες και ένωση κεφαλαγορών. Τον... Θα τον ευχαριστήσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα από κοντά. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ επειδή ο πρόεδρος Γιούγκερ αποφάσισε το χαρτοφυλάκιο αυτό, το επιτόπου Χιλ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαίου στον αντιπρόεδρο Μπρόφσκης. Εσείς ε, ε, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, αμέσως μετά εκφράσατε την ε, διαθεσιμότητά σας να έρθετε εδώ να συναντηθείτε με την Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προσωπικά αλλά και οι συντονιστέ, θελήσαμε να σας καλέσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Το χαρτοφυλάκιο που καλύπτετε εσείς, που καλύπτει την Ένωση Κεφαλαγορών, την Τραπεζική Ένωση, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και γενικότερα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι ένα χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικό τη στιγμή που προσπαθούμε ακόμα να διορθώσουμε τα προβλήματα και να διορθώσουμε έναν τομέα ο οποίος είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης όλος ιδιαίτερος. Ως μέρος λοιπόν της προπαρασκευαστικής εργασίας σας έστειλα γραπτές ερωτήσεις από τους συντονιστές της Επιτροπής μας. Τις γραπτές σας απαντήσεις τις μοιράσαμε στους βουλευτές. Η γραμματεία έχει ετοιμάσει και σε χαρτί τις απαντήσεις αυτές. Υπάρχουν βέβαια στα αγγλικά μόνο, δεν είχαμε καιρό να τις μεταφράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως που μας απαντήσατε τόσο γρήγορα στις ερωτήσεις μας. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στην ακρόασή μας με τους συνήθεις κανόνες. Δηλαδή εσείς θα έχετε το λόγο για μια εισαγωγική παρουσίαση 10-15 λεπτά και μετά 5 λεπτά ο καθένας, 2 λεπτά ερώτηση και 3 λεπτά απάντηση για τον κάθε ευρωβουλευτή. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω εδώ σήμερα και να συζητήσω μαζί σας. Με λύπησε η απόφαση της 23ης Ιουνίου του δημοψηφίσματος, αλλά πρέπει να τη σεβαστούμε. Και ο Επίτροπος Χίλ αποφάσισε να παραιτεθεί. Σέβομαι την απόφαση αυτή, παρόλο που με λυπή που χάνω ένα τόσο καλό συνάδελφο. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στα όσα έκανε ο Επίτροπο Χιλ και στην καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μα. Το εύχομαι βέβαια ότι καλύτερο για το μέλλον. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε σημαντικούς καιρούς γεμάτους προκλήσεις. Οι διαδικασίες, οι χρηματοπιστωτικές αλλά και οι πολιτικές χρειάζονται σημαντικές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, ασφάλεια, μεταναστευτικό κλπ. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από κάθε αλλαγή στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αμένο Βασίλειο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμα στο μέλλον πώς θα είναι οι σχέσεις μας αυτές. Ελπίζουμε όμως, ελπίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να είναι στενός εταίρος μας. Και προς το παρόν παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Συγχρόνως 27 χώρες μέλη υπόλοιπε ξεκαθάρισαν ότι οτιδήποτε διευθετήσεις γίνουν στο μέλλον το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια τρίτη χώρα και βάσει αυτού θα πρέπει να δούμε τι υποχρεώσει και τα δικαιώματά τη. Η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά σημαίνει ότι πρέπει να δεχτεί όλε τι ε, ελευθερίε του Ηνωμένο Βασίλειο για τα αγαθά, του ανθρώπου, τα κεφάλαια και τι υπηρεσίε. Δεν μπορεί να επιλέγει ό,τι θέλει και να αφήνει τα υπόλοιπα. Ο πρόεδρο Γιούγκερ λοιπόν μου ζήτησε να αναλάβω εγώ τις, την ευθύνη του χαρτοφυλακίου για, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και ένωση κεφαλαιογορών από τον Ιούλιο. Θα ήθελα αυτό να έχει γίνει κάτω από διαφορετικέ συνθήκε, καλύτερε συνθήκε, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πρόκληση αυτή για μένα και την αναλαμβάνω. Ω αντιπρόεδρο επίτροπο, ήδη ήμουν αρμόδιο για το συντονισμό του χαρτοφυλακίου αυτού, για την Τραπεζική Ένωση για την ευάθυνση στην ΟΝΕ και για τα χρηματοπιστωτικά. Έτσι λοιπόν, από την εμπειρία μου ως ε, Ευρωβουλευτής, γιατί ήμουν Ευρωβουλευτής πριν γίνω Επίτροπος, έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. Επιτρέψα μου τώρα να σας πω πώς βλέπω εγώ το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι να ενισχύσει την οικονομία, να τη χρηματοδοτήσει και να προστατεύσει και την κοινωνική οικονομία. Έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση των startups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορέσει αποτελεσματικά να διαχειριστεί τα οικονομικά του, την εκπαίδευση και να προστατευτεί από το χάος. Αποτέλεσμα της κρίσης είναι ότι ενισχύσαμε την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σήμερα είναι πιο ισχυρός από ό,τι πριν από την κρίση. Η οικονομία μας βελτιώνεται. Οι τράπεζές μας είναι περισσότερο ισχυρές και με περισσότερα κεφάλαια. Όμως, οι επενδυτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Προχωρώντας λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε μια καλή ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια στέρεα εποπτική βάση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η ρύθμιση για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της αλυσίδας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ανοιχτό σε νέες εξελίξεις στην κοινωνία, στην τεχνολογία, με μια καλή διάρθρωση του τομέα κάθε φορά που αυτό χρειάζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια ένωση μια εσωτερική αγορα για όλες τις χώρες μέλη και με κοινό νόμισμα για πολλές από τις χώρες μέλη. Αυτό είναι και το δικό μου χαρτοφυλάκιο που είμαι αρμόδιο για το ευρώ, οπότε συντονίζω και το ευρωπαϊκό εξάμεινο που συμμετέχουν όλε οι χώρες μέλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ και να γίνει πιο δυνατή, να στέκεται καλύτερα. Γι' αυτό και πρέπει όλες οι χώρες να είναι ισχυρές. Τα πρόσφατα γεγονότα βέβαια τάραξαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα παντού. Έχει να κάνει με την εφαρμογή ή μη της, των κανόνων της ΟΝΕ σε όλους τους τομείς, σε όλες τις πλευρές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είτε πρόκειται για εγγύησεις, είτε για οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιέζουμε όλες τις χώρες μέλη ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες. Και πρέπει επίσης να περάσουμε και σε ένα νέο επίπεδο ε, διακυβέρνησης και να διασφαλίσουμε ότι τους επόμενους μήνες οι προτάσεις μας για το TLAC και το MREL θα προχωρήσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Και χαίρομαι που οι Υπουργοί έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν ένα νέο, ένα νέο backstop Πρέπει επίσης να προχωρήσει το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων. Αποτελεί μέρος βέβαια ενός ευρύτερου σχεδίου προκειμένου να βαθύνουμε περισσότερο στην Οικονομική Ένωση. Όλα αυτά βρίσκονται τώρα στα χέρια των δύο συνομοθετών. Γι' αυτό και τους επόμενους μήνες και εβδομάδες θα συζητήσω πολύ μαζί σας, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο φυσικός εταίρος μας και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν χρειαζόμαστε διακυβερνητική συμφωνία για να ολοκληρώσουμε. Το ΕΝΤΙΣ πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με άλλα μέτρα για να μειωθούν οι κίνδυνοι στο τραπεζικό τομέα. Οι προτάσεις μας για το LAC και το CRD θα είναι έτοιμες πριν από τα τέλη της χρονιάς. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε προδιαγραφές να ισχύουν και να εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συνεργαστούμε με την Βασιλεία και θα συντονίσουμε και τις ρυθμίσεις αυτές. Περιμένουμε βέβαια τη δική σας συνεισφορά στις συζητήσεις για τέτοια ζητήματα. Όσον αφορά τώρα την Κεφαλαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο του Επιτρόπου Χίλ για να οικοδομήσουμε την Ένωση Κεφαλαγορών και συνεργαζόμαστε με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν πολύ για αυτό το τομέα. Πρέπει η Ένωση Κεφαλαιογορών να ολοκληρωθεί ακόμα πιο γρήγορα, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση κάποιες επιχειρήσεις να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή η ΟΝΕ για να μπορεί να απορροφά καλύτερα όλους τους κραδασμούς. Του χρόνου θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε μετά τις τωρινές προτάσεις και δράσεις και να δούμε τι παρετέρω μπορούμε να κάνουμε. Πάντως πρέπει να επικεντρωθούμε σε συμφωνία πάνω στις ήδη υπάρχουσες προτάσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας για να έχουμε ένα καθεστώς το οποίο να λειτουργεί καλύτερα, να είναι πιο φθηνό για όλες τις επιχειρήσεις και να λειτουργεί πιο εύκολα βάσει αυτού η αγορά. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για να προχωρήσουμε πάνω στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με διαφάνεια και βάση ξεκάθαρων προτύπων. Οι καταναλωτέ πρέπει να έχουν περισσότερη επιλογή όσον αφορά τις δημοσιονομικές υπηρεσίες. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Και τώρα αναλύουμε τις απαντήσεις μετά από τη διαβούλευση που έγινε βάσει τη πράσινη βίβλου μας. Και θέλουμε να καταλήξουμε το φθινόπωρο σε προτάσει σε συμπεράσματα. Το FinTech τώρα είναι επίση ένα τομέα πάνω στον οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους την βιωσιμότητα ε, στις δικές τους επενδυτικές πολιτικές. Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε στην πολιτική μας βάση αποδείξεων, ώστε να στηρίζουν όλες μας οι δράσεις στην ανάπτυξη. Προχωρήσαμε και στο λεγόμενο Call for Evidence, την πρόσκληση για υποβολή στοιχείων, και τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει θα τα χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που παραμένουν στο σύστημα. Όσον αφορά τώρα τους CCP, τους συμβαλόμενους, και εκεί πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να είναι πιο ισχυροί για να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση. Για να ολοκληρώσω, πολλές προκλήσεις παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Είναι μια βαριά ατζέντα, πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αλλά προσβλέπω σε συνεργασία, καλή συνεργασία μαζί σας για να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Ο Μπούρχαρ Μπάρτς, πρώτος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα καταρχάς να απευθυνθώ ε, στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τον ευχαριστήσω που βρίσκεται σήμερα εδώ. Ε, μετά από την απόφαση να δοθεί σε εσά το, το χαρτοφυλάκιο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ήρθαμε σε επαφή μαζί σας ε, και αμέσως απο, αποφασίσατε να έρθετε στην Επιτροπή μας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι από το ΕΛΚ. Επίσης, ε, μιλάω ε, για το γεγονός ότι εσείς εκτιμάτε αυτό το σώμα καθώς το γνωρίζετε ως Ευρωβουλευτής. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη δουλειά μας χωρίς εσάς. Ε, το είπε ήδη ο Πρόεδρος ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε προσωπικά για τη δουλειά που έχει γίνει ως τώρα. Με τον κύριο Ντομπρόφσκης λοιπόν ως αντιπρόεδρο ε, πρέπει να μιλήσουμε για και έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά για όλα τα στοιχεία του ευρώ. Έχετε τώρα και την Τραπεζική Ένωση στο χαρτόφυλάκι σας και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε ασχοληθεί με ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολύ πιο πολύπλοκες, πιο λεπτομερείς. Εσείς λοιπόν έχετε πιο πολλές ρυθμιστικές ικανότητες. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας, πρέπει τακτικά να μπορούμε να ε, εποπτεύουμε και τις μεγάλες ε, τράπεζες αλλά και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το Call for Evidence που αναφέρατε ήταν αποτέλεσμα αυτής της επιτροπής, αιτήματος αυτής της επιτροπής να γίνει μια ενδελεχής μελέτη. Ε, τώρα λοιπόν η δική σας ε, αρμοδιότητα ε, έχει να κάνει με αυτό το call for evidence που πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό με ενίσχυση της αναλογικότητας γιατί πρέπει πάντοτε τακτικά να κοιτάζουμε την αναλογικότητα και να διασφαλίσουμε ότι τα στάνταρτ, οι ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, δεν ε, παραβιάζονται και γίνεται σεβαστή και η βούληση των νομοθετών. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Βάλτσε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση για το Call for Evidence. Ακριβώς αυτό είναι και ο στόχος της πρόσκλησης για την συλλογή ε, στοιχείων είναι ακριβώς αυτό ε, που θα έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο στο ρυθμιστικό μας χαρτοφυλάκιο, στη ρυθμιστική ατζέντα. Ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε είναι να έχουμε γρήγορα ε, βελτίωση επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε συγκεκριμένα αιτήματα για call for evidence να τα αναλύσουμε ένα προς ένα και αναλάβουμε δράση όταν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν το call for evidence είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την επίτευξη ενός καλύτερου ρυθμιστικού πλαισίου. Υπήρξε μια έντονη ε, αντίδραση και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις, αλληλοεπικαλύψεις ε, και οι ασυμβατότητες μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών ε, εργαλείων. Γενικά το θέμα αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της μεταρρύθμισης του συστήματος του πλαισίου διακυβέρνησης που έχει τεθεί σε ισχύ τα τελευταία χρόνια. Τώρα για την ανάλυση των αντιδράσεων φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις ομάδες που αναδύονται. Η μία είναι αυτή που εξετάζει το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα αναλογική η νομοθεσία μας, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση που υπάρχει διαθέσιμη για την πραγματική οικονομία σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις η συμμόρφωση τελικά οδηγεί σε αλληλοεπικαλύψεις, ασυμβατότητες και άλλα τέτοια προβλήματα. Περιμένουμε λοιπόν την ανάλυση και μέσα στους επόμενους μήνες και εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε καλύτερα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε υπερβάσεις Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Τίποτα. Όπως και πολλοί και εμείς ε, θέλουμε κρίμα που έφυγε ο κύριος Χιλ. Νομίζουμε ωστόσο ότι η αλλαγή του χαρτοφυλακίου τροποποιεί την αρχιτεκτονική που αρχικά είχε διαμορφώσει ο πρόεδρο τη επιτροπή ε, και θεσμικά και πολιτικά. Τούτο ωστόσο δεν ε, είναι ούτε δική σας ευθύνη ούτε της ακράσεως. Μία ερώτηση για το τι πιστεύετε σχετικά με τη σημασία της συγχώνευσης μετά τον και του ε, χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης και του Λόγκο Stock Exchange. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα αντιμετωπίσετε είναι το θέμα του διαβατηρίου διότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται αυτού του διαβατηρίου μπορεί να παράσχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος μέλος η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, ούτως διότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, ούτως ώστε να μπορέσει να, προσφέρει, να προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές. Πώς θα εξασφαλίσει η Κομισιόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρεί τις υποχρεώσεις του ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίω από την περίοδο τώρα, από τη τωρινή στιγμή και ιδίω μέχρι το κλείσιμο των ε, διαπραγματεύσεων αποσχόλησης. Τέλος, η Επιτροπή σε συνδυασμό με τις SMA, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, έχει την πρόθεση να εποπτεύει τις δυνατότητες κατάχρησης της αγοράς που συνδέονται με δραστηριότητες που διεξάγουν ιδίω. Ε, ε, φορείς της εκστρατείας του Brexit που μπορεί να εκμεταλλευτούν την ταραχή στην αγορά που προέκυψε από το δημοψήφισμα πριν ή μετά. Okay. So, um, thank you uh, very much for those... Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κάμποσες. Πρώτον, ο αντίκτυπος του δημοψηφίσματος στη Βρετανία στις σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις πιθανές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τούτο σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τι μοντέλο σχέσεων θα έχει τελικά η Βρετανία με την Ένωση. Γενικά δύο εναλλακτικέ υπάρχουν. Η μία να συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι μέλος της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και ένα δεύτερο εκτός. Προφανώς γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά περιλαμβάνει και υποχρεώσεις ε, τέσσερις ελευθερίες αλλά και χρηματοοικονομική συμβολή στην Ένωση και σεβασμός προς, την, προς το νομικό πλαίσιο που λειτουργεί στην Ένωση. Γνωρίζουμε ότι το θέμα του, της διαβατηριοποίησης συνδέεται με την συμμετοχή μιας χώρας στην εσωτερική αγορά της Ένωσης. Αν μείνει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο στην η ερώτησή μου είναι τι γίνεται πριν το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων και το καθεστώς της Βρετανίας. Πριν, τώρα δηλαδή, η Βρετανία συνεχίζει να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό. Θα συνεχίσει να είναι σε αυτή τη θέση έως ότου ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 της συνθήκης και ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Μέχρι τότε, για δύο χρόνια τουλάχιστον ακόμα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το σεμβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι που όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης πρέπει να σέβονται. Στην περίπτωση αυτή, ίσως και η, όπως τόνισε και η κανονιστική αρχή της Βρετανίας, θα πρέπει να συνεχίσει η Βρετανία να σέβεται όλη την νομοθεσία της Ένωσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Όσο είναι μέλος της Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και όλους τους κανονισμούς της Ένωσης. Για το ερώτημα της κατάχρησης αγοράς. Θα έλεγα ότι έχουμε ένα αρκετά καλό νομικό πλαίσιο και στην οδηγία και στον κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς. Οι κανονιστικές αρχές έχουν μια σειρά εργαλείων στη διάθεσή τους για την καταπολέμηση καταχρήσεων στην αγορά και να επιβάλλουν κυρώσεις στους υπεύθυνου αν διαπιστωθούν τέτοιες πράξεις. London Stock Exchange και η Φραγκφούρτη. Τώρα για το χρηματιστήριο του Λονδίνου, επαναλαμβάνω, όσο η Βρετανία παραμένει πλήρες μέλος της Ένωσης, δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις, νομικά τουλάχιστον. Υπάρχει ένα θέμα ευθύνων, αρμοδιοτήτων για την αγορά, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει στο τέλος, αν θα μείνει ή όχι η Βρετανία σαν μέλος της, κοινή, της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήλθατε. Κρίμα που σας καλούμε εδώ λόγω του ότι έφυγε ο κύριος Χίλ και λόγω του αποτελέσματος στη Βρετανία είναι κάτι που δεν θα ήθελα προσωπικά. Αλλά τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που υπογραμμίσετε ότι η, Ένωση, ότι η Βρετανία παραμένει πλήρες μέλος της Ένωσης ε, καθοδόν προ την διαπραγματεύση. Ξέρετε ότι οι συντηρητικοί υποστήριζαν ε, τον Λόρδο Χιλ και την ικανότητά του να, να εξισορροπεί και το call for evidence και μια ε, προοδευτική ε, ημερήσια διάταξη CMU. Εκτιμώ το ότι ήδη ε, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό στην πρώτη ερώτηση, αλλά θα ήταν χρήσιμο να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει η πρόσκληση για υποβολή ε, αποδεκτικών στοιχείων στο επίπεδο 2, σε περιπτώσεις MIFID για παράδειγμα, όταν ζητούμε αποδεκτικά στοιχεία, ενώ ο χρόνος που χρειάζεται για την ενώ απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας πριν παρασκευθούν αυτά τα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ισορροπούν τα νέα νομοθετικά κείμενα και τα υφιστάμενα νομοθετικά κείμενα. Πώς θα εξισορροπείτε η προσέγγιση σας για τον ρόλο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και χρηματοοικονομικής, ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και ίσως να μπορούσατε να μας πείτε πώς θα χρησιμοποιήσετε τη μεθοδολογία αυτής της, προσ, της πρόσκλησης υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Όπως ξέρετε, στην Επιτροπή θέσαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα σε ένα σταθερό και υγιές χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι το σύνολο του ε, ε, ότι χρειαζόταν μια αναμόρφωση του χρηματοοικονομικού νομοθετικού κειμένου μετά την κρίση για να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που είχαμε στο χρηματοοικονομικό τομέα. Και μάλιστα οι πρόσφατες αναταραχές στην αγορά σε σχέση με το Βρετανικό Δημοψήφισμα υπογράμμισαν εκ νέου την ανάγκη να έχεις μια, έναν ανθεκτικό χρηματοοικονομικό τομέα και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο Ίσως λοιπόν δεν είναι αντιφατικές οι δύο προσεγγίσεις. Θέλουμε σταθερό και υγιές χρηματοοικονομικό σύστημα ως προϋπόθεση για να υποστηρίξουμε την οικονομία μας. Τώρα για την εξισορρόπηση που αναφέρατε και να έχουμε μια φιλόδοξη ε, ημερήσια ε, και, ε, και ένα φιλόδοξο θεματολόγιο και να καταλάβουμε τι έχουμε δημιουργήσει. Αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει ήδη πολύ ακόμα νομοθετική δουλειά. Μια σειρά προτάσεων συζητούνται ήδη στην Επιτροπή σας. Θα, έρθουμε, θα έρθουν κι άλλες, ανεφερορισμένες, στην αναθεώρηση του κανονισμού κεφαλαιακών απεπτήσεων, της οδηγίας, της διεθνείς απαιτήσει για το TLAC που θα πρέπει να προσαρμοστούν στη δική μας MLAC μια σειρά άλλων δηλαδή νομοθετικών κειμένων. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο δημιουργήθηκε και κάπως ad hoc, σαν μια απάντηση στην κρίση. Αυτή η πρόσκληση λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων που αναλύεται αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να σταθούμε και να δούμε πώς είναι συνολικά το πλαίσιο, αν υπάρχουν ασυνέπειες, επικαλύψεις και πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα χωρίς πολύ, δημοσιο... πολύ ε, διοικητικό βάρος. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την ε, νομοθεσία βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Προφανώς σεβόμαστε την αρχή αυτή, το υπογράμμισε και εισαγωγικά. Όταν αποφασίζουμε για σημαντικά ζητήματα που ενδεχομένως έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις και για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να στηριχθούμε σε αποδεικτικά δεδομένα και αυτή την προσέγγιση θα συνεχίσω να την ακολουθώ όπως έκανε και μέχρι τώρα ο Λόρδος Χιλ. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους του Άλντε. Χαιρετίζω την ποιότητα του έργου του Επιτρόπου Χίλ και το θάρρος του για την απόφαση που πήρε που τον τιμά απόλυτα. Στην ακρόαση αυτή τώρα, ας πάρουμε κάποια απόσταση σε σχέση με τους φακέλους που έχουμε την τάση να εξετάζουμε χωριστά. Θα σα ρωτήσω στο τέλο για την Επιτροπή τη Βασιλεία. Προηγουμένω όμω θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω εσεί που πάτε διακοπέ, κύριε Επίτροπε, αλλά ελάτε μαζί μου στην Aix-en-Provence και να μου εξηγήσετε πώ εγώ μπορώ να πω εκεί στου απλού ανθρώπου, ακόμα και αν νομικά έχετε απόλυτα δίκιο, και δεν έχω καθόλου επιθετικότητα κατά των Βρετανών, αλλά ρωτάω, εκτός των χώρων που εδώ γνωρίζουμε καλά, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε απλούς πολίτες ότι για ένα χρονικό διάστημα που δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι αυτό, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, δεν είμαστε σε μεταβατική περίοδο, είμαστε σε ένα περίοδο αγνώστου διάρκειας, οι Βρετανοί εδώ θα ψηφίζουν κείμενα που δεν θα τους αφορούν, θα έχουμε ίσως έναν νέο επίτροπο που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκι εγώ, εγώ θα πω ας ε, κάνουμε μια εκστρατεία γιατί θα είναι πάρα πολύ περίεργο το να έχουμε εδώ πέρα έναν Βρετανό επίτροπο. Θα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος αν μη τι άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε... Ε, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, με τους Βρετανούς δηλαδή, ώστε νομικά να είμαστε εντάξει απέναντι στους Βρετανούς, που να διακανονίζουν όσο γίνεται καλύτερα την κατάσταση, αλλά συγχρόνως να μας επιτρέπει να αμυνθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των λαϊκιστών που θα επωφεληθούν για να πούνε ότι εμείς είμαστε εντελώς ξεκομμένοι από την πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή επιπλέον απόλυτη εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Λοιπόν, πείτε μου, πέρα από το να επαναλαμβάνετε το νομικό δόγμα, τι έχετε να μου πείτε. Γιατί ακριβώς η Επιτροπή που μας λέει ότι είναι πολιτική δεν είναι δυνατόν μόνο νομικά επιχειρήματα να μας προτείνει. Έρχομαι τώρα και σε κάτι άλλο. Βρεθήκαμε με τη Μαντελβό και άλλους, ετοιμάσαμε την έκθεση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, στα standard settings, εκεί δηλαδή που ε, κανονίζονται οι λογιστικές προδιαγραφές. Πέρα από αυτήν την μικρή έκθεση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θεωρήσει καλύτερα τις σχέσεις μας κυρίως με την Επιτροπή της Βασιλείας. Κάποιες αποφάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας θα υιοθετηθούν σύντομα. Εσείς τι θα κάνετε αν το αποτέλεσμα των εργασιών ε, αυτών που είναι σημαντικές βέβαια γενικά δεν ανταποκρίνονται στα όσα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Απάντηση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, για την κατάσταση μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλες οι χώρες μέλη πρέπει να σέβονται τη συνθήκη. Και υπάρχουν διατάξεις στη συνθήκη. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη όπου μια χώρα μέλος σκοπεύει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο ο ευρωπαϊκός θεσμός δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σεβαστούμε τη συνθήκη. Και η συνθήκη είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι η χώρα μέλος πρέπει να ενεργοποιήσει το άρθρο 50. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν είναι απεριόριστη η περίοδος, γιατί άπαξ και ενεργοποιηθεί το 50, έχουμε δύο χρόνια για τη διαπραγμάτευση. Αυτό προβλέπει η συνθήκη. Δεύτερον, η Προεδρία των Θεσμικών Οργάνων ζήτησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει στην κοινοποίηση ώστε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 χωρίς καθυστέρηση. Και όντως αυτή η περίοδος αβεβαιότητας, συμφωνώ μαζί σας, ότι είναι σημειογόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάμε από το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει την κοινοποίηση αυτή χωρίς καθυστέρηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τηρούμε τις συνθήκε. Τώρα όσον αφορά τη Βασιλεία και τις διεθνεί εργασίες. Όπως είπα και εισαγωγικά, καλωσορίζουμε τη δικιά σας ε, συνεισφορά με την έκθεση πρωτοβουλίας που εκπονήσατε όσον αφορά το έργο για τη συνεισφορά, IMF, Βασιλεία κλπ. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν να μιλάει με μία φωνή. Γιατί τότε μπορούμε να επηρεάσουμε καλύτερα το έργο των διεθνών αυτών φόρα. Και το δεύτερο είναι ο συντονισμός στο IMF, στο Δουνουτού δηλαδή, έχουμε κάνει πρόταση για καλύτερη εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ. Τι θα γίνει τώρα αν τα αποτελέσματα της Επιτροπής Βασιλείας δεν ευθυγραμμίζονται με την ειδική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, αν μιλάμε με μία φωνή μπορούμε καλύτερα να πειράσουμε τα πράγματα. Και δεύτερον, το είπα με το TLAC. Όταν το εφαρμόζουμε, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε με φύ τρόπο, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις δικές μας ρυθμίσεις και με τις απαιτήσεις του MREL. Πρέπει να γίνεται ώστε να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έληξε ο χρόνος σας, ε, ε, κυρία Γκουλάρη, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, επόμενος. Ε, κύριος Φάμπιο Νταμάφσκι. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Ντομπρόφσκης. Θα ήθελα επειδή εδώ ε, η συζήτηση για τον Brexit ε, μεν παίζει μεγάλο ρόλο, εμείς ως ε, Ευρωπαίοι είμαστε τώρα αντιμέτωποι και με μια κατάσταση η οποία μοιάζει με νηπιαγωγείο. Ε, στην οποία μπροστά το Brexit μοιάζει είναι Είναι η, κρίση, η κρίση ε, για τις Ιταλικές τράπεζες. Ε, έχετε έρθει σε επαφή με την Ιταλική κυβέρνηση. Πώς ε, θα διαχειριστείτε τα υφιστάμενα ε, προβλήματα, ειδικά ως προς το θέμα της ιδιοκτησίας ε, και των πιστωτών που θα πρέπει να λάβουν, αναλάβουν τις ευθύνες τους, πώς θα προστατέψουμε τους μικρούς επενδυτές και αποταμιευτές, ε, διότι εσείς πάντοτε ήσασταν υπέρ του Συμφώνου Ανάπτυξης, εμείς αντιθέτως πάντοτε το επικρίναμε στην ομάδα μου και Φαίνεται ότι η Ιταλία πρέπει να δώσει έως και 2,5% του ΑΕΠ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των τραπεζών, οπότε δεν θα μπορεί να τηρήσει το σύμφωνο. Επίσης, σύμφωνα με μία μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών, ε, φαίνεται ότι η Deutsche Bank είναι η τρίτη τράπεζα για την παγκόσμια σταθερότητα. Μιλήσατε για την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών, μιλήσατε για τις πιστοτικές ε, δραστηριότητες. Πώς θα προχωρήσετε λοιπόν με αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι σωστό και βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη ε, ιδρύματα όπως η Deutsche Bank ε, που αυτή επηρεάζει την παγκόσμια σταθερότητα να τα πιέζουμε. Επίσης ο κύριος Χίλ είχε αφήσει, έχει αφήσει πίσω του ένα πολύ ενδιαφέρον ε, χαρτοφυλάκιο, δεν θα, σας, δεν θα βαρεθείτε, όμως ε, ίσως ε, είναι υπερβάλλον να έχουμε έναν τέτοιο ε, επίτροπο για αυτό το θέμα, είχατε πει κάποτε, ήταν ο κύριος Χίλ ε, ε περιτός και τι θα κάνετε εσείς με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Κοιτάξτε, ήταν πολλές ερωτήσεις. Για το πρώτο ερώτημα, για τις Ιταλικές τράπεζες, να πω ότι όντως υπάρχουν πολλές ε, δυσκολίες στον Ιταλικό τομέα, τον τραπεζικό. Έχουμε μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε μεγάλο ποσοστό και έχουμε και μη ε, και έλλειψη κερδοφορίας της τράπεζας. Ε, Επίσης μειώνονται και οι τιμές των μετοχών. Όμως αυτό δεν είναι μια νέα εξέλιξη, είναι κάτι που ισχύει από την αρχή του έτους. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το έχουμε ήδη τονίσει στις ειδικές συστάσεις που έχουμε κάνει προς την Ιταλία. Ε, έχουμε πει ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί όπως ας πούμε ένα συγκεκριμένο ε, το Atlanta ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την τιτλοποίηση αυτών των δανείων και φαίνεται ότι οι Ιταλικές αρχές ε, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και είναι και έτοιμες να δράσουν εάν χρειάζεται. Μετά, για την ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών. Ε, σας, άκουσα, σας ρώτησα πώς συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, κύριε πίτροπε. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εξαρτάται και από τις Ιταλικές αρχές, ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν. Ήδη έχουν εφαρμοστεί κάποια πράγματα πάντοτε σε στενή συνεννόηση με τις Ιταλικές αρχές. Αλλά να περάσω λίγο γρήγορα και στα άλλα ερωτήματα για την μεταρρυθμίση της δομής των τραπεζών. Ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση έχει κολλήσει προς το παρόν. Δεν προχωράει. Κάποιες από τις ανησυχίες που προέκυψαν ήταν ε, πώς για παράδειγμα θα συνεχίσουν οι τράπεζες να να παρέχουν ε, συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες όπως market making, η αναλογικότητα Αυτά είναι οι ανησυχίες. Ε, άρα, ε, εγώ θέλω να έρθω σε επαφή με τους εισηγητές ε, και τους σκιώδεις για να μπορούμε να δούμε μαζί πώς θα προχωρήσουμε. η πρόταση ήθελε ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσει το θέμα των πολύ μεγάλων τραπεζών που δεν μπορούμε να αντέξουμε την κατάρρευσή τους. Αυτό το πρόβλημα παραμένει. Για, το, ε, για την επόμενη πρόκληση που αναφέρετε στην ερώτησή σας, να πω ότι θα την αναλάβω. Πάντοτε συντόνιζα την εργασία αυτή ως αντιπρόεδρος ούτως ή άλλως. Δεν είναι οι ευθύνε μου καινούριε λοιπόν και καταλαβαίνετε ότι στην Επιτροπή ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά μέλη που είναι υπεύθυνα για διάφορες γενικές διευθύνσεις και μπορούν με επιτυχία να αντιμετωπίσουν τέτοιες προκλήσεις. Εντάξει, είναι επιπλέον δουλειά, αλλά είμαι έτοιμος να την αναλάβω. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Σβέν Γκίγκολ. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να μιλήσω λίγο για τον τρόπο που έχουμε στην ΕΚΟΝ, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, να αντιμετωπίζουμε τις ε, διαπραγματεύσεις που θα επέλθουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Να πω ξεκάθαρα και στη Σιλβή ότι πραγματικά ε, η περασμένη εβδομάδα ήταν μια λυπηρή συγκυρία. Ο τρόπος, το στυλ με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πρέπει να είναι φιλικός, να μην υπάρχει καμία εχθρικότητα, καμία διάθεση εκδίκησης ο τόνος που εσείς χρησιμοποιήσατε λέει ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ίδιοι κανόνες, ίδιες υποχρεώσεις. Όσο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στα χέρια του και στα χέρια των υπόλοιπων μελών της κοινή αγοράς φυσικά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ως προς τις υποχρεώσεις. Όποιος είναι στην κοινή αγορά πρέπει να σέβεται όλες τις υποχρεώσεις όπως ας πούμε την ελεύθερη κίνηση των προσώπων και των αγαθών αλλά και τις πληρωμές στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα λέμε με έναν τόνο φιλικό και είναι σωστό να έχουμε το σωστό τόνο στις μελλοντικέ μας σχέσεις με τους πολίτες των Ηνωμένου Βασιλείου και ιδιαίτερα των νέων που θέλουν να έχουν ένα μέλλον στην Ευρώπη. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα για σας κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς με ανησύχησαν ειδικά ε, τα, οι απαντήσεις που δώσατε για το RTS 21, για τα ε, όρια της, θέση, τα, ε, της θέσης, τα position limits. Ε, είπατε ότι υπάρχει ανησυχία από το Κοινοβούλιο. Να σας πω ότι πολλοί πολίτες ανησυχούν για το θέμα. Είστε έτοιμοι να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Θέλετε να έρθετε να συναντήσετε εμένα και την ομάδα διαπραγμάτευσης για το MIFID πριν πάρετε την απόφασή σας για το RTS 21. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, για την αναπτυσσόμενη αγορά των πράσινης χρηματοδότησης, ποια μέτρα θα πάρετε για να υποστηρίξετε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα, να περάσει η οικονομία μας σε μια μετάβαση προς την οικολογία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, για τις ερωτήσεις μάλλον. Ε, πρώτα, να απαντήσω για το RTS 21 και τα position limits, τα όρια θέσεις. Σημεριζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρα τους στόχους αυτού του στάνταρ, δηλαδή με αυτό το πρότυπο θέλουμε να μειώσουμε την κερδοσκοπία ως προς τα βασικά αγαθά Τελεία. Ε, γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητήσαμε από την ΕΣΜΑ να επανακαταθέσει την πρόταση και να επανέλθει με ένα βελτιωμένο στάνταρτ για τα όρια θέσης, ένα βελτιωμένο πρότυπο στην αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΣΜΑ είδαμε ότι υπάρχουν περισσότερες διαφοροποιήσεις ε, έχουμε χαμηλότερα όρια, λιγότερο, λιγότερα ρευστά ε, συμβόλαια και επίσης όρια όπου ε, τα τρόφιμα είναι το παραδοτέο αγαθό είναι σε ένα ε, όριο του 2% του εφοδιασμού. Αυτό που είπα και στη γραπτή μου απάντηση είναι ότι έχω την αντίποση, εντύπωση ότι ε, φαίνεται να ικανοποιούνται οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Δηλαδή πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Ε, βέβαια το θέμα θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πεδίο. Επίσης, για το δεύτερο ερώτημα που ε, θέσατε σχετικά με την πράσινη οικονομία. Η πράσινη χρηματοδότηση και η οικονομία είναι ζητήματα που αφήνουν μεγάλο περιθώριο δράσης. Χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, στρατηγική για αυτό το θέμα. Ε, αυτό επίσης συνάδει και με τη δουλειά μας στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο FSB και στο G20. Θέλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε πρακτικά τις διάφορες εφαρμογές. Ας πούμε την προσέγγιση που έχουμε για τις επαγγελματικές συντάξεις, πώς θα δράσουμε και σε άλλους τομείς, ε, αν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση για παράδειγμα στο CRR και στο CRD ε, και επίσης ε, είμαι έτοιμος να συζητήσω και άλλους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Μάρκο Τζάνι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ακρόαση. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, εν γέννη για το μέλλον της Τραπεζικής Ένωσης. Ε, η κρίση που βιώνουν ορισμένα κράτη και η Ιταλία μεταξύ άλλων αφορά στον τραπεζικό τομέα που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για την δομή της Τραπεζικής Ένωσης. Είναι η δομή αυτή ικανή να δώσει σταθερότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρώπης, όπως είχε ως αρχικό στόχο Έχουμε έναν πυλώνα, την ενιαία εποπτεία που είναι άνισος πυλώνας γιατί ασχολείται μόνο με κάποιους ε, κινδύνους που εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς των τραπεζών αλλά αγνοεί τους μεγαλύτερους. Με ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι όπως έλεγε ο συνάδελφος Ντεμάζη μια τράπεζα όπως η Deutsche Bank με βάση τα stress test του SSM φαίνεται ότι είναι μια ε, λίγο επικίνδυνη η τράπεζα και μετά έχετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι η τράπεζα αυτή είναι ένας από τους ισχυρότερους συστημικούς κινδύνους στην Ευρώπη. Κάτι δεν στέκει. Έχουμε ένα σύστημα εξυγίανσης που φαίνεται ότι αντί να σταθεροποιεί το χρηματοοικονομικό σύστημα το θέτει σε κίνδυνο. Οι εθνικές αρχές που εφάρμοσαν με μερικό ή πλήρη τρόπο είδαν τις επιπτώσεις και στην αγορά. Αρκεί να δείτε την απόδοση στον, ε, στα χρηματιστήρια από, το, από τον Ιανουάριο του 2016 του τραπεζικού κλάδου και των τραπεζών σε κάποιες χώρες. Γίνεται ό,τι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εφαρμόσουν οδηγία αυτή, διότι αν την εφαρμόσουν θα δημιουργήσουν τεράστια ταραχή στον ε, τραπεζικό τομέα, ιδίω αν εφαρμοστεί αυτό σε μεγάλες τράπεζες, συστημικές τράπεζες. Κατόπιν υπάρχει ένας τρίτο πυλώνας που φυσικά δεν θα υλοποιηθεί ποτέ ή αν υλοποιηθεί θα είναι κάτι που δεν θα χρησιμοποιησει ιδιαίτερα για να γίνει ασφαλές το ευρωπαϊκό σύστημα. Οι σκέψεις του λοιπόν μετά από κάποιο χρόνο για, για, το, για το κατά πόσον ε, είναι δυνατή να λειτουργήσει η Τραπεζική Ένωση. Δεύτερον, securitization συχνά η, κεντρική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας λέει ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι η έλευση ρευστότητα, αλλά ζήτηση. Είναι, είναι σωστή η λύση, μια περαιτέρω χρηματοποίηση της πραγματική οικονομίας όπως προκύπτει από την Banking Union. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις πάλι. Πρώτον, Τραπεζική Ένωση. Εγώ όπως σας είπα θα συνεχίσω να ασχολούμαι και να δουλεύω για την Τραπεζική Ένωση με επιπλέον προτάσεις την ε, εποπτική παράμετρο όπως ε, υπογραμμίστηκε και θα ε, δουλέψουμε και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων που είναι το, ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Κατόπιν, για την λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού SSM και τις διάφορες διαστάσεις των επιμέρους κινδύνων. Εγώ θεωρώ ότι η κίνδυνη της μη εξυπηρέτησης και του trading είναι σοβαρή κίνδυνη, Όπως ξέρετε ωστόσο, ο υπεύθυνο για την εποπτεία είναι ο SSM και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλύπτεται τούτο από τις ρυθμίσεις για την εξαρτησία της. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένα συγκεκριμένες αποφάσεις των υποπτικών αρχών. Τώρα, για την ε, securitization, τιτλοποίηση. Αυτό έχει σαν στόχο να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση στην οικονομία. Εμεί θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόταση για ένα ενιαίο σύστημα, ομοιόμορφο σύστημα τίτλοποίηση είναι θετικό γιατί επιτρέπει στι τράπεζε να περάσουν τα, τα, τα στοιχεία του σε πιθανού επενδυτέ, ούτω ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία προ όφελο τη τελευταία. Αναφερθήκατε στην πλευρά τη ζήτηση τη οικονομία όντω. Ο χρηματοοικονομικός τομέας δεν μπορεί να λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Έχουμε ευρύτερα, ευρύτερη θεματολογία στα μακροοικονομικά, έχουμε προτεραιότητες για την διευκόλυνση των επενδύσεων, για την, τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις και την προσπάθεια τόνωσης τη ζήτηση στην οικονομία, ιδίως στις χώρες εκείνες ε, που έχουν δημοσιονομικό χώρο γι' αυτό. Εκεί αυτό είναι, αυτό είναι κομμάτι και της ημερήσια διάταξής μας. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τον καλημερίζω. Τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και τώρα ε, που αναλάβατε και το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Χίλ έχετε πολύ μεγάλες αρμοδιότητες. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε πολύ καλή συνεργασία και στο εξής. Πριν από αυτήν εδώ την ε, ακρόαση, ήδη απαντήσατε κάποιες ε, ερωτήσεις και κάνατε και μία ε, τοποθέτηση αρχικά για το σύστημα εξασφάλισης των επενδύσεων. Το ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούνιο μίλησε εντατικά για το θέμα αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα και μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Το είπατε βέβαια ήδη ότι είστε κατά αυτής της συμφωνίας ε, και ε, συγκεκριμένα έχει να κάνει αυτό με τη μείωση του ρίσκου και με την ε, οδηγία για την εξυγίανση που έχει δύο διαστάσεις αφενός να Έχουμε την αποσύνδεση των τραπεζών από τα κράτη, έχουμε το θέμα της Ιταλίας για παράδειγμα, έχουμε και άλλα κράτη όπου ε, λειτουργεί καλά ε, το ταμιευτήριο ας πούμε όπως στην Αυστρία. Έχουμε δηλαδή ε, ένα σύστημα στην Ευρώπη στο οποίο λειτουργεί η εξασφάλιση γενικά και έχουμε μια γενικότερη μείωση του ρίσκου. Όμως ε, θέλω να δούμε πώς η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα έχουν τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια και πώς θα διασφαλίσουμε και την πιθανότητα να υπάρξει ε, κατάρρευση μιας τράπεζας. Ε, υπάρχει μια μελέτη η οποία θα πρέπει να γίνει σε σχέση με τη διασφάλιση του κόστους. Επίσης, άλλη μια ερώτηση που έχει να κάνει με την επιρροή των ε, ε, rating ε, των ιδρυμάτων, δηλαδή οργανισμούς χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης. δεν μπορούμε πάντοτε να βασιζόμαστε σε, αυτές, σε αυτούς θα πρέπει ε, πολλές φορές ε, να ε, ρυθμιστικά να μην παρεκκλίνουμε και θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας. Απάντηση. Πάλι πολλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το έντις. Όπως είπα και πριν, σκοπεύω να συνεχίσω το έργο που έχει ήδη αρχίσει για το ΕΝΤΙΣ, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εξασφάλισης Καταθέσεων. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι στα χέρια των συνομοθετών το ζήτημα. Το ΕΚΟΦΗΝ έχει ήδη καθορίσει το χάρτη πορείας του για το πώς να προχωρήσουμε και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τη Σλοβακική Προεδρία προκειμένου να αρχίσει το τεχνικό έργο για το φάκελο αυτό και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια το οποίο ε, δουλεύει πάνω σε αυτό. Υπάρχει ήδη ένα έγγραφο το οποίο εκπονείται. Οπότε είμαι έτοιμος και εγώ να συνεργαστώ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για τις διάφορες πτυχές. Πρώτον, όσον αφορά το εθνικό σύστημα εγγύσεων. Η πρόταση έντις διευκρινίζει ότι μόνον οι χώρες μέλη οι οποίες καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους υπό το πλαίσιο της οδηγίας για την εγγύηση καταθέσεων θα υποφεληθούν από το έντις. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει μια κατάσταση για χώρες οι οποίες δεν έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις των της οδηγίας με εθνικό σύστημα γύρισης καταθέσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, πόρους από το έντις σε βάρος άλλων χωρών. Άρα, το 0,8% ε, πρέπει τελικά να επιτευχθεί. Έπειτα αναφερθήκατε στην Αυστρία, σε αποταμιευτήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν θα καθορίσουμε τις συνεισφορές βάσει κινδύνου. Και ήδη κάτι έχει γίνει. Σκοπός μας δεν είναι να αυξήσουμε συνολικά το βάρος για όλες τις τράπεζες. Το 0,8% θα παραμείνει ο στόχος μας για τις καταθέσεις όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα. Τώρα για την μείωση κινδύνου. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι ο επιμερισμός κινδύνου και η μείωση του κινδύνου πρέπει να γίνουν εκ παραλίλου. Και έχουμε εξετάσει διάφορες προτάσεις που μας έφτασαν όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου. Όσον αφορά τώρα τις οικονομικές υποχρώσεις βάσει του Μπέιλιν. Το Ταμείο Εξυγίανσης μπορείτε να φτάσετε μόνο εφόσον υπάρχει ένα ποσοστό bail-in. Είναι πράγματα τα οποία διευκρινίζονται στο MREL. Οπότε ποιες είναι οι οικονομικές υποχρώσεις εξαρτάται από αυτό και με ποια σειρά. Τώρα για την αξιολόγηση κόστους. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια εκτίμηση αντικτύπου πλήρης ήδη από το 2010, όπου εξετάσαμε διαφορετικούς τρόπους πανευρωπαϊκού συστήματος εξασφάλισης καταθέσεων. Είμαστε έτοιμοι πάντως να συνεργαστούμε πιο στενά και να εκτιμήσουμε παρετέρου διάφορα στοιχεία τα οποία θα ήθελε το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο για να αποφασίσουν. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και παρετέρω ανάλυση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. του όρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σήμερα το πρωί στο ξεκίνημα της ε, παρεμβασής αναφερθήκατε στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ε, λόγω της μετανάστευσης, ασφάλειας, της αβεβαιότητας και των κινδύνων που η διακοπή της, Ευρωπαϊ... της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ενωπήσης στην Αγγλία δημιουργεί. Αν δείτε τις σημερινές ε, φωτογραφίες θα δείτε ότι χτες επέστρεψαν στην Ιταλία οι ισορροί ε, εννέα Ιταλών που δολοφονήθηκαν από την Ισλαμική Τρομοκρατία στο Μπαγκραντές. Οι σελίδες των εφημερίδων είναι γεμάτες από πληροφορίε για την τράπεζα Monte dei Paschi di Siena που έχασε 30% της αξίας της σε λίγες μέρες. Η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε για να δούμε πώς θα χειριστούμε μια πιθανή μελλοντική κρίση εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της εταιρείας είναι σημαντικό πρόβλημα. Η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πλαίσιο μας παρέχει εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοια κατάσταση. Θέλω να καταλάβω αν τα κενά που βλέπουμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μήπως επιδεινώνουν την κατάσταση. Τέλη Ιουλίου θα γίνουν τα νέα stress test της, Ευρωπαϊ... της EBA που θα ασχοληθούν εκ νέου κυρίως με τα με εξυπηρετούμενα δάνεια και όχι με τον σύνθετο χαρακτήρα των ε, ισολογισμών των τραπεζών που περιλαμβάνουν παράγωγα και δημιουργούν σοβαρού κινδύνου, Όπω είναι, είπαν και οι συνάδελφοι, και το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, οι κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματο στην Ιταλία δεν έρχονται από τα δάνεια, αλλά από την, ε, τα προβλήματα που δημιουργεί η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα. Την ερώτηση, παρακαλώ, λέει ο πρόεδρο. Η ερώτηση είναι αυτή. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η Ευρώπη, η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει γρήγορη δράση. Τι πιστεύετε για την χρήση της ευελιξίας που προβλέπει το, η οδηγία για το BRD, άρθρο 2.4 Δέλτα που ζητά να υπάρξει επίγουσα παρέμβαση για να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι την κάλυψα ήδη όσον αφορά τις Ιταλικές τράπεζες. Βέβαια δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω η ιδιαίτερη κατάσταση για την συγκεκριμένη τράπεζα. Πάντως, διάφορα βήματα όσον αφορά το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα έχουν ήδη αναλυφθεί και αυτό σε στενή συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές. Έπειτα, ρωτήσατε για το BRRD, την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών. Πράγματι, όταν εφαρμόζουμε τους κανόνες, εφαρμόζουμε όλες τις διατάξεις των κανόνων, ανάλογα με τις προϋποθέσεις. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται για να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία προβλέπει η BRRT. Αλλά είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις αυτές που πρέπει, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι τράπεζες. Να ανταποκρίνονται στις κεφαλαϊκές απαιτήσει βάσης και μετά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα η προληπτική διαχείριση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα μέτρα και αν οι προποθέσεις καλύπτονται μπορούν και να εφαρμοστούν. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρεται στους κανόνες και είναι βέβαια αρμοδιότητα του Επιτροπού Βεστάγκερ αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε εφικτές λύσεις συνολικά ως Επιτροπή. Μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει σε διάφορες περιπτώσεις για το θέμα της στήριξης ρευστότητα και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα να εργαζόμαστε. Τώρα για τις διάφορες πτυχές κινδύνου ήδη είπα ότι πράγματι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορους κινδύνους, είτε εμπορικούς, είτε διάσωσης. Πάντως, ειδικέ λύσεις πρέπει να υιοθετούνται από τις εποπτικές αρχές κάθε φορά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον προκατοχό σας και να σας πω ότι μας καθισκάζει όταν αναλαμβάνετε εσείς το χαρτοφυλάκιό του. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό μας δίνει αρκετές εγγύσεις. Μία και μόνο ερώτηση έχω προς εσάς η πραγματική δοκιμή για το αν έχουμε πραγματικά μια τραπεζική ένωση. Έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στις τράπεζες της Βόρειας Ευρώπης, κατά πόσο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στη Νότια Ευρώπη, όπου υπάρχουν προγράμματα αλλά οι τράπεζες πολλές φορές βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Σήμερα δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Όχι εξαιτία του πρωτογενούς ή του παράγωγου δικαίου, αλλά γιατί οι εθνικοί ρυθμιστές στις χώρες του Βορρά φροντίζουν οι αποταμιεύσεις τους, οι καλές αποταμιεύσεις τους, να μην τεθούν σε κίνδυνο σε επενδύσεις σε χώρες που θεωρούνται λιγότερο σοβαρές. Στον ε, προκάτοχό σας το είχα επίση ρωτήσει, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ πιστικά. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή. Έχει να κάνει με τον κατακαιρματισμό της χρηματοπιστωτικής φελεκής αγοράς και με την τάση την οποία έχουμε διαπιστώσει από την αρχή της κρίσης όπου υπάρχει μερικώς τουλάχιστον επαναθνικοποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων όπου το χρήμα δεν κυκλοφορεί τόσο πολύ διασυνοριακά. Πράγματι, ένας από τους στόχους του έργου μας είναι ακριβώς αυτό με την κεφαλαϊκή αγορά, να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό αυτών και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μια πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες όσον αφορά όλες τις πτυχές της κελεφικής αγοράς. Εσείς στις τράπεζες αναφερθήκατε, αλλά υπάρχουν στοιχεία εδώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρώτα απ' όλα η αναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου, εποπτικός μηχανισμός που ήδη προβλέπεται και δουλειά προκειμένου να μην υπάρχουν πια τα διάφορα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με την πράσινη βίβλο μας στο χρηματοπιστωτικό τομέα να δούμε πώς δηλαδή θα προωθήσουμε τις λιανικές ε, υπηρεσίες διασυνοριακά. Παραμένουν βέβαια και εμπόδια που είναι γλωσσικά ή νοοτροπίας. Υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα προστασίας των καταναλωτών που και αυτά πρέπει να ε, τα δούμε. Διαφορετικά επίσης συστήματα όσον αφορά την αφαιρεγκαιότητα πώς αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα στις διάφορες χώρες. Και υπάρχει το FinTech και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ώστε να υπάρξει διαφορά στις δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα διασυνοριακά. Υπάρχουν διαφορετικοί πολλοί τρόποι δηλαδή για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και φροντίζουμε γι' αυτό στην πράσινη βίβλο μας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η αναθεώρηση της κεφαλαϊκής αγοράς θα είναι μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσουμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση και να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό τον κατακαιρματισμό. Ευχαριστούμε. Ολτάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πιο, ακόμα πιο απαιτητικό φαίνεται να γίνει το χαρτοφυλάκιο και τον Ντομπρόφσκι. Έχω τρει ερωτήσει που θα σα ζητούσα να απαντήσετε και να λάβετε θέση. Διότι μερικέ φορέ ε, τις χάνονται. Πρώτον, Ένωση Κεφαλαιογορών, Capital Market Union, ως πρόγραμμα δράσης. Προφανώς θα υπάρξει συνέχεια από πλευρά σας, αλλά οι συνθήκες άλλαξαν υπάρχει πλέον το Brexit. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το τέλος της ε, Ένωσης Κεφαλαγορών που και ο λόγος ε, που είχε πάρει την, ε, το χαρτοφυλάκι αυτό ένας Βρετανός ήταν, ήταν συγκεκριμένος. Άλλοι λένε το ανάποδο, ότι τώρα μπορεί να, να εμβαθύνει η Ένωση την αγορά. Δεύτερον, πρόσκληση υποβολή στοιχείων, call for evidence. Η Ένωση λέει ότι ναι, είναι χρήσιμο αυτό, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, ασυνέπειες και τις επικαλύψεις. Αν δείτε όμως ε, τη θέση του Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι η θέση μας είναι ευρύτερη. Δεν μιλάμε μόνο για ασυνέπειες, αλλά για να ζητάμε από την Επιτροπή να εξετάσει τα πιθανά, ε, τα πιθανά ζητήματα. Υπήρχε το θέμα της υπερ ε, νομοθέτησης. Μετά, τιτλοποίηση. Είχαμε μια μακρά συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, που ασχολήθηκε περισσότερο με τα διδάγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε από τη χρηματοοικονομική κρίση. Και σε μία από αυτές τις συζητήσεις ο κύριος Χίλ εδώ, υποστήριζονται στην προσέγγιση αυτή. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια αγορά όχι μόνο στις καλές εποχές αλλά και τις κακές που θα μπορεί να κάνει το χρηματοοικονομικό τομέα όχι μόνο σταθερό και ισχυρό αλλά και με δυνατότητα να παρέχει ρευστότητα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ένωση κεφαλαγορών και επιπτώσεις του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Όπως είπα εισαγωγικά, ενισχύεται η ανάγκη της Ένωσης Κεφαλαγορών, ιδίως όταν ο κίνδυνος είναι η μεγαλύτερη αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη να μετακινηθεί εκτός Ένωσης. Αυτές που θα κερδίσουν από την, από την αγορά κεφαλαγορών, άλλωστε είναι οι χώρες με, μικρότερες, με λιγότερο ισχυρές αγορές κεφαλαίου. Θα ήθελα να προωθήσω το θέμα αυτό και δεν συμφωνώ με την θέση σας ότι το δημοψήφισμα οδηγεί στο τέλος της αγοράς ε, της Ένωσης Κεφαλαγορών στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε για όλη την Ένωση με θετικά και για την ΟΝΕ. Τώρα, το call for evidence. Και εδώ υπάρχουν κενά. είναι η αξιολόγηση μας είναι συνοδική, καλύπτει όλες τις διαστάσεις μεταξύ των οποίων και τα κενά και τις ε, τρύπε. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα υπόλοιπα κενά στον κανονισμό των χρηματαγορών, Φερρυπίν, την ρύθμιση των ή ένα πλαίσιο εξυγένσης CCP αν θέλουμε να καλύψουμε και κινδύνους στις δομές αυτές. Τα διδάγματα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η τίτλοποίηση όντως ε, έχει κακή φήμη λόγω της κρίσης των subprime στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Να δει η Ευρώπη προϊόντα που είναι σύνθετα, και, και, και δάνεια που γίνονται με μόνο σκοπό να απολυθούν σε άλλους. Η κατάσταση της τιτλοποίησης, της ωστόσο στην Ευρώπη και της ΕΠΑ είναι διαφορετικές. Ακόμα και στην περίοδο της κρίσης, τα προϊόντα τιτλοποίησης στην Ένωση που είχαν πάρει τριπλό α, ε, ε, βρέθηκαν σε πτώχευσαν μόνο σε 0,01% των περιπτώσεων, ενώ στην, ε, στις ΗΠΑ αυτό αφορούσε το 16%. Τώρα, εμείς θα υποβάλουμε μια πρόταση για ένα απλό, ομοιόμορφο και τυποποιημένο σύστημα τιτλοποίησης που θα μειώσει τον κίνδυνο των τιτλοποιήσεων και θα επιτρέψει στους καταναλωτές να καταλαβαίνουν ευκολότερα τον κίνδυνο των πιθανών κινδύνων. Ξέρουμε ότι και οι εποπτικές και οι κεντρικές αρχές ε, υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας και η Επιτροπή της Βασιλείας. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί είναι τι πρέπει να γίνει για να γίνει η πρόταση όσο καλύτερη γίνεται ούτω ώστε να λειτουργήσει η τιτλοποίηση και σε καλές και σε κακές χρονικές στιγμές. Ευχαριστώ. Ο Πάμπλο Ζάλμπα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει. Τιτλοποιήσει. Σε συνέχεια αυτών που αναφέρθηκαν και ω υπεύθυνο εισηγητή ε, για την κεφαλογορά. Ποια είναι η άποψή σα για την πρότασή μου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εράχηση των ε, ε, εμφάσεων που θέλει να δώσω. Ε, θέλουμε να φύγει η εξωτερική μέθοδος προ όφελο της εσωτερικής αγοράς. Ποια είναι η άποψή σα σχετικά. Δεύτερον, αξιοπιστία και ε, σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά και της Ευρωζώνης συνολικά. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, ότι στις, οι νέες σας ευθύνες δεν, σε εμποδίσουν να δουλέψετε για να πετύχετε το στόχο της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και στο χρηματοοικονομικό σύστημα ε, και ακόμη περισσότερο μετά το Brexit που είχε έναν αντίκτυπο και όχι θετικό θα έλεγα στην αξιοπιστία εμείς θεωρούμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι να αναζητήσουμε και να ανακτήσουμε αυτή την πληγωμένη αξιοπιστία. Η ερώτησή μου είναι τι τι δυνατότητε, μάλλον τι, τι αξιοπιστία δίνει το να επιβάλλεται κυρώσει σε μια χώρα που έχει ανάπτυξη και που μπορεί να δώσει ε, αρνητικές επιπτώσεις στην σταθερότητα τη Ευρωζώνη και του χρηματοοικονομικού συστήματος. Μήπω αυτό είναι ένα λάθο μήνυμα ιδίω σε μια στιγμή που πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση. Μια χώρα που αναπτύσσεται, που κάνει μεταρρυθμίσεις, είναι μια χώρα που θα πρέπει να υποστεί κυρώσεις από την οπτική της αξιοπιστίας επαναλαμβάνω και τη σημασία που η αξιοπιστία θα έχει στην, στο χρηματοοικονομικό σύστημα και την Ευρωζώνη. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά και ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Φυσικά η η ακρόση αυτή έχει να κάνει με το νέο χαρτοφυλόκιο του κυρίου Ντομπρόφσκης, αλλά μπορείτε να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις αν θέλετε. Θα ξεκινήσω απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση, γιατί φοβάμαι ότι από την μετάφραση δεν κατάλαβα την πρώτη. Ίσως μπορείτε να μου την επαναλάβετε λίγο γρήγορα μετά. Για το δεύτερο ερώτημα. Φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας, πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ε, ανάπτυξη και τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται. Αυτό είναι που κάνουμε. Αν δείτε τις προτεραιότητες ε, που έχουμε σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής θα δείτε ότι είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον ε, εξυγχρονισμό των οικονομιών μας και η συνέχιση και ενίσχυση των ε, υπεύθυνων πολιτικών σε ε, δημοσιονομικό επίπεδο. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την κατάσταση που υπάρχει στις περισσότερες χώρες, το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος να κρατά όμοιρο την ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν ε, να είμαστε... Έχουμε λοιπόν ε, ε, πολλή δουλειά να κάνουμε. Ταυτόχρονα, αν δούμε συνολικά τη δημοσιονομική θέση, ήδη βρισκόμαστε συνολικά σε μία ε, κατάσταση στην ζώνη του ευρώ που υπάρχει μια επέκταση. Ο νομαστικός προϋπολογισμός ε, το, το ισοζύγιο μειώνεται αλλά διαρθρωτικά αυξάνεται. Συνολικά λοιπόν τα κράτη-μέλη είναι σε υπερβολικά ελλείμματα τα οποία ε, οδηγούν σε μια ανάγκη για συνέχιση της προσπάθειας προσαρμογής. Όσον αφορά το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, να πω ότι φυσικά το εφαρμόζουμε με έναν ε, εύλογο τρόπο, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό που έκανε ως τώρα η Ισπανία και φυσικά και η Πορτογαλία, σε επίπεδο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Βέβαια δεν μπορώ να σχολιάσω τις αποφάσεις της Κομισιόν πριν ληφθούν, όμως συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Μοσκοβιστή πολύ στενά σε αυτό το θέμα. Το είπε χθε δημοσίως και αυτός ότι δεν μπορούμε να σχολιάζουμε αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί ακόμα αλλά φυσικά ε, συγχαίρουμε τις χώρες αυτές και λαμβάνουμε υπόψη τις προσπάθειες που έχουν κάνει για μεταρρυθμίσεις και προσαρμογή και για την εφαρμογή του συμφώνου. Για την πρώτη ερώτηση να ζητήσω να την επαναλάβετε. Δεν έχουμε χρόνο, ε, θα τα συζητήσετε όλα αυτά, είμαι σίγουρος, ε, με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκι σε άλλη ευκαιρία. Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, που ήρθατε σήμερα εδώ. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω, παρακαλώ, σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Η πρώτη έχει να κάνει με τη δημιουργία του backstop. Τι μορφή θα έχει. Μπορείτε ως Αντιπρόεδρος, ως Επίτροπος, αρμόδιος τώρα και για την Ένωση Κεφαλαιογορών να μας πείτε πώς θα σχεδιαστεί αυτό το backstop. Δεύτερον, θέλω να μάθω για το ΕΝΤΙΣ, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εξασφάλισης Καταθέσεων. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει για την ανάγκη να εργαστούμε εκ για την ανάπτυξη του ΕΝΤΙΣ και για επιπλέον μέτρα μείωσης του κινδύνου. Αυτό το έργο που λέμε να πάει εκ παραλίλου δεν ορίζεται καλά. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από τη μια θα έχουμε το EDIS και από την άλλη μεριά θα έχουμε το TLAC, το MREL, το δημόσιο χρέος κλπ. Δηλαδή το EDIS σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα ε, δεν ξέρω πού θα σταματήσει η διαπραγμάτευση για το έντις. Έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο λοιπόν για την μείωση του κινδύνου, αλλά δεν νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το ίδιο όταν λέμε ότι πρέπει να δουλέψουμε συγχρόνως και για το έντις αλλά και για άλλα συνοδευτικά μέτρα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αυτό το έργο εκ παραλίλου. για αυτά που είπε πριν και ο κύριος Γουαλτιέρη όσον αφορά την ακραίωση αυτή. Απλώς θέλω να προτείνω ότι τώρα που υπάρχουν αβεβαιότητες για το ευρώ θα πρέπει να υποφεληθούμε από κάθε είδους ευελιξίας όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και να αποφύγουμε κυρώσεις σε χώρες για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ισπανίας έκανε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις ε, λαϊκίστικου τύπου, αλλά αυτό το θέμα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί συζητάμε τώρα για την ίδια την εξοπιστία της Ευρωζώνης και το μέλλον του ευρώ. Οπότε πριν πάρουμε μέτρα ιδιαίτερα αυστηρά, επιθετικά, θα έπρεπε να το σκεφτούμε ξανά και ξανά. Απάντηση. Πρώτον, όσον αφορά το κοινό backstop. Οι υπουργοί, και αυτό είναι το θετικό, συμφώνησαν να δουλέψουν για αυτό το κοινό backstop. Οπότε θα αρχίσουμε το τεχνικό έργο πολύ σύντομα. Για τον ακριβή ρυθμό και την κατεύθυνση που θα πάρει το έργο αυτό, ως Επιτροπή θέλουμε να διευκολύνουμε τη συμφωνία αυτή, οπότε είμαστε ανοιχτοί. Εξετάζουμε διαφορετικούς τρόπους για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του κοινού backstop, οπότε θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε έγκαιρα. Δεύτερον, για το έντις και για το τι εννοούμε με τον επιμερισμό κινδύνου και την μείωση του κινδύνου και τα σχετικά μέτρα, πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά παράλληλα. Εμείς το είπαμε σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν υποβάλαμε νομοθετική πρόταση για το έντις και είπαμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και για την μείωση κινδύνου. Αν όμως δείτε την νομοθετική μας πρόταση για το έντις, το έντις δεν αποτελεί προϋπόθεση για το ένα ή το άλλο μέτρο. Έδι, ήδη έχει πάει στους συνομοθέτες οι οποίοι και το συζητούν. Βεβαίω σημειώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές χώρες και διαφορετικά σημεία αναφοράς. Και το είπατε και εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι πρέπει πρώτα να βασιστούμε στη μείωση του κινδύνου, το δημόσιο χρέος, άλλοι λένε με το έντις μετά, άλλοι λένε το έντις τώρα και η μείωση κινδύνου μπορεί να περιμένει. Ε, συνεπώς πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Γιατί ακριβώ αυτό το θέμα του επιμερισμένου κινδύνου και της μείωσης του κινδύνου είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε και ήδη τα σχέδια κειμένων δείχνουν να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επί όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητα και την ευελιξία εφαρμογή του. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πήρε ήδη από τον Ιανουάριο του 2015 ήταν μια ανακοίνωση για την καλή χρήση της ευελιξίας στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οπότε έχω ήδη απαντήσει και απάντησα και σε προηγούμενο συνάδελφο και είπα ότι θα κοιτάξουμε τις διάφορες προϋποθέσεις και με τον Επίτροπο Μοσχοβησή θα συνεργαστούμε στενά για να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. Ευχαριστώ. Κρίστιαν Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Θα μιλήσω αγγλικά σήμερα. Ξέρουμε ότι έχετε ένα με, μεγάλο παρελθόν ε, ε, καλής ας πούμε απόδοσης ως Πρωθυπουργό ε, στη χώρα σας. Ε, ε, έχετε εφαρμόσει γρήγορες μεταρρυθμίσεις που μετά από ένα χρόνο οδήγησαν σε ανάπτυξη. Επίσης μπήκατε στην Ευρωζώνη. Ελπίζω οι ικανότητέ σας για τη διαχείριση μιας κρίσης να μην χρειαστούν στην τρέχουσα κατάσταση όπως χρειάστηκε στη Λετωνία πριν από πολλά χρόνια. Τώρα, για την συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, το Brexit δημιουργεί πολλές ε, αναταραχές στην αγορά. Ξέρουμε ότι όταν ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 θα υπάρχουν δύο χρόνια περιθώριο, όμως δεν γνωρίζουμε πότε θα ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι ο μεγάλος άγνωστος. Τώρα, οι ψηφοφόροι μας γενικά ε, καταλαβαίνετε ότι θέλουν να έχουν μια δουλειά, θέλουν να έχουν ένα μισθό για να πληρώνουν τα έξοδά τους και για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις και ένας τραπεζικός τομέας που θα χρηματοδοτεί αυτές τις επενδύσεις. Άρα το ερώτημά μου, υπό το φως όλων αυτών που συμβαίνουν και της αβεβαιότητας που υφίσταται παρά το τι επιθυμούμε εμείς θα μπορέσει να αντισταθεί ο ευρωπαϊκός ε, τραπεζικός τομέας. Υπάρχουν άμεση κίνδυνοι που βλέπετε λόγω της αβεβαιότητας. Χρειάζεται να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα εμείς ειδικά ως νομοθέτες για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Είναι γενικό το ερώτημά μου. Απάντηση. Για τους κινδύνους στην αγορά μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Είδαμε ότι οι αγορές αντέδρασαν ηχηρά. Υπήρξε μια απότομη πτώση στα χρηματιστήρια, ειδικά στα κεφάλαια που, έχουν, που θεωρούνται πιο ε, επικίνδυνα αυτά που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις δραστηριότητες εκεί. Υπήρξαν άμεσες απώλειες αμέσως μετά το δημοψήφισμα, σε μεγάλο βαθμό λοιπόν, σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, έπεσαν, ε, ε, ε αυξήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, αυξήθηκε η τιμή του χρυσού, και έπεσαν οι τιμές των μετοχών και των βασικών αγαθών. Και στην Ευρωζώνη είδαμε κινητικότητα γύρω από κάποιες τράπεζες. Η κατάσταση βέβαια κατά κάποιο τρόπο έχει σταθεροποιηθεί έκτοτε και έχουν κάπως ανακάμψει οι αγορές όσον αφορά στις απώλειες που υπέστησαν αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Οι κεντρικές τράπεζες, η έκτη η Τράπεζα της Αγγλίας ήταν πολύ καλά προετοιμασμένες και έδειξαν ετοιμότητα για να ε, αναλάβουν υποστηρικτική δράση ε, εφόσον καταστεί απαραίτητη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Γενικά βέβαια η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε τα γεγονότα και να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε γέρος εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ευχαριστούμε. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης, είναι πολύ καλό που είστε εδώ και με χαρά μου άκουσα ότι σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε το θέμα ε, της, των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλες και δεν πρέπει να αποτύχουν ε, επανενεργοποιώντας ε, τα ζητήματα που έχουν μείνει αδρανή. τώρα πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε την ε, έκθεση πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας οριζόντιας tax force. Αναφέρατε στη γραπτή σας απάντηση ότι ο Λόρδος Χιλ είδε, ήδη είχε φτιάξει μια εσωτερική ομάδα δράσης για το FinTech, όμως ε, ε, αυτό έχει να κάνει με τεχνολογία και έξυπνα συμβόλαια τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα και γι' αυτό χρειάζεται μια οριζόντια ομάδα δράσης. Άρα αναρωτιέμαι αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή τη σύσταση. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι πιο γενική. Με ανησυχεί το Brexit, βλέπουμε μια νέα σειρά φορολογικού ανταγωνισμού από τα διάφορα ε, χρηματοπιστωτικά κέντρα εις βάρος των ε, πολιτών. Το City στο Λονδίνο ε, εξασθενεί λόγω του δημοψηφίσματος και αρχίζουν να υπάρχουν πιέσεις για λιγότερη φορολογία και τα χρηματοπιστωτικά κέντρα στο Παρίσι, τη Φραγκφούρτη, το Λουξεμβούργο ελπίζουν να προσελκύσουν περισσότερες δραστηριότητες και κάποια έχουν ανακοινώσει ήδη φορολογικά πλεονεκτήματα για να το επιτύχουν. Το ερώτημά μου είναι πώς θα σταματήσετε αυτό αυτή την καθοδική πορεία ε, προς ε, μια, ένα τέτοιο ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, για τις τεχνολογίες καταρχάς, ε, της blockchain, να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία με πολύ μεγάλο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια πιο προσεκτική ρυθμιστική προσέγγιση γιατί αυτή η τεχνολογία πρέπει να αναπτυχθεί και να δείξει το δυναμικό της. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα εικονικά νομίσματα για παράδειγμα, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να εξετάσουμε σχετικά με τα εικονικά νομίσματα στο σχέδιο δράσης, ε, ας πούμε, για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αξιολογούμε και προτείνουμε να επιτραπεί στις αρμόδιες αρχές να έχουν μια εποπτεία αυτών των ε, συναλλαγών και να μπορούν να παράγουν ε, αυτά τα στοιχεία που συγκεκριμένα μπορεί να χρειάζονται κάθε φορά. Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει κάτι τέτοιο να παρακολουθείς και να παράγει στοιχεία για κάθε ε, συναλλαγή ανά πάσα στιγμή, απλώ πρέπει να βρούμε την κατάλληλη υποδομή. Ανέφερα επίσης στι γραπτές μου απαντήσεις ότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργείται μια εσωτερική ομάδα δράσης στην Κομισιόν για το FinTech και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να βρούμε έναν τρόπο για να δημιουργήσουμε την οριζόντια task force που αναφέρατε, γιατί πρόκειται για νέα τεχνολογία και χρειάζεται πραγματικά να δούμε τα διάφορα ε, στοιχεία αυτής της οικονομικής τεχνολογίας, της FinTech. Δεν ε, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά, έχει και εφαρμογές στον τομέα των επικοινωνιών και ούτω καθεξής. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να εργαστούμε από αυτό. Μετά, για το δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα, διότι εάν δείτε το πνεύμα της εργασίας μας ε, στη φορολογία, ας πούμε, η βάση του ΟΣΑ για την ε, διάβρωση της βάσης και την μετατόπιση των κερδών μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Άρα στις προτάσεις της Κομισιόν και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στην αρμοδιότητα του κυρίου Μοσκοβισή ε, προσπαθούμε να έχουμε μία προσέγγιση βάσει της οποίας τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα. Να μην μεταφέρονται κάπου αλλού για φορολογικούς λόγους. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το εντομετωπίσουμε αυτό. Υπάρχουν ε, οι αρχές της αποφυγής διπλής φορολογίας που μας βοηθούν να το κάνουμε αυτό Ας πούμε, θέλουμε την ε, πραγματική και αποτελεσματική φορολογία ε, βάσει αυτών των αρχών και ένα κράτος μπορεί να δράσει αν εισόδημα σε άλλη χώρα δεν έχει τύχη της ε, σωστής φορολόγησης. Επίσης υπάρχουν οι κανόνες για τις κρανικές ενισχύσεις είναι κάποιες αποφάσεις φορολογικές, ας πούμε, που δίνουν πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτές ε, μπορεί να θεωρηθούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Πρόκειται λοιπόν να χρειαστεί και αυτό το θέμα να το παρακολουθήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε και έχουν ήδη υπάρξει πολλές ε, πρωτοβουλίες. Φυσικά αξίζει να παρατηρήσουμε ότι από ευρωπαϊκή άποψη η φορολογία είναι ένας σύνθετος τομέας γιατί όλα τα ζητήματα φορολογίας απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Γνωρίζοντας όμως αυτούς τους περιορισμούς, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε και να έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε... ευχαριστώ Πρόεδρε. Φτάνουμε στο τέλος της ανταλλαγής αυτής απόψεων, οπότε επιτρέψτε μου να μην ρωτήσω για το έντις εγώ, γιατί πολλοί ρώτησαν μέχρι τώρα για το έντις. Θέλω όμως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον Αντιπρόεδρο, που μπόρεσε και ήρθε τόσο νωρίς σήμερα το πρωί να μας δει. Πολλές ερωτήσεις έγιναν και για το δημοψήφισμα, το Brexit. Πολλές από αυτές φυσικά έχουν άμεση σχέση με, το, με την Επιτροπή μας Οικονομικών Υποθέσεων και εννοείται ότι όλους μας απασχολεί το πόσο αποτελεσματικά θα μπορούμε να δουλέψουμε. Άλλες ερωτήσεις όμως σχετικά με το Brexit δεν έχουν να κάνουν ε, με την Οικονομική Επιτροπή θα μπορούσαν να τεθούν οπουδήποτε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σε οποιοδήποτε άλλον, γιατί είχαν να κάνουν ε, με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 κτλ. Δεν έχουν να κάνουν με τα οικονομικά ζητήματα και τη δικιά μας δουλειά εδώ. Πάντως η επίπτωση του Brexit, αν αποχωρούσε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη θα την έβλεπαν πολύ σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ταυτίζονταν αυτά τα δύο. Επικίνδυνο, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη, που μπορεί να προσθεθούν στην Ευρωζώνη, αλλά εσείς πώς θα αποφύγετε αυτές τις διακρίσεις ε, όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση μεταξύ των χωρών που είναι στην Ευρωζώνη και εκείνων που δυνητικά θα συμμετάσχουν κάποια στιγμή. Αυτό θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και δεν το ρωτήσαμε ακόμα, οπότε πολύ θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό και σε οτιδήποτε άλλο δεν συζητήσαμε ενδεχομένω μέχρι τώρα στην ακρόαση αυτή. Απάντηση. Για την Ευρωζώνη, αυτούς που συμμετέχουν και αυτούς που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. Γίνονται διάφορα θέλουμε. Εμβάθυνση όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με την έκθεση των πέντε προέδρων έχουμε προχωρήσει και εμείς ε, στα διάφορα στάδια. Έχουμε εφαρμόσει το πρώτο στάδιο και δουλεύουμε πάνω στο δεύτερο στάδιο και θα υπάρξει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από αυτού πολύ σύντομα. Τώρα έχουμε τονίσει από την αρχή ότι όλες οι πρωτοβουλίες θα είναι ανοιχτές και απόλυτα διαφανείς και απέναντι στις χώρες που δεν συμμετέχουν στο ευρώ. Και θα σχεδιαστούν οι πρωτοβουλίες με τέτοιο τρόπο ώστε οι χώρες μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη να μπορέσουν να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες αυτούς, αυτές. Από εκεί και πέρα. Όλα τα ζητήματα που συζητάμε ε, συζητιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ό,τι συζητάμε για την ΟΝΕ δεν γίνονται σε βάρος των χωρών που συμμετέχουν στην ε, εσωτερική αγορά. Και αυτή η προσέγγιση πρέπει να συνεχιστεί. Όταν συζητάμε για την Τραπεζική Ένωση, βλέπουμε ότι de facto αυτή η Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει τις χώρες ευρώ, αλλά είναι ανοιχτή και σε χώρες εκτός ευρωζώνης, εφόσον αποφασίσουν να συμμετάσχουν και αυτή η δυνατότητα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και σε οποιαδήποτε μελλοντική μας νομοθετική δράση. Προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ακρόαση αυτή και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που δεχτήκατε να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας. Υποθέτω ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι. Τώρα οι συντονιστές κάπως ε, άτυπα θα συνεδριάσουμε απλώς για να διαπιστώσουμε τι βγήκε από αυτήν την ακρόαση την οποία εγώ εκτίμησα όλους Σε Ευχαριστούμε πολύ, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Ε, ε, και εγώ σας ευχαριστώ και προσβλέπω και εγώ στη συνεργασία μαζί σας για όλους αυτούς τους σημαντικούς φακέρους που συζητήσαμε σήμερα.